την ε, διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στην Κίνα. Έχετε το λόγο κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, η προστασία δεδομένων είναι θεμελιώδη δικαίωμα στην Ένωση και ισχύει και όταν μεταφέρονται προσωπικά στοιχεία εκτός Ένωσης. Το Κοινοβούλιο αυτό παίζει βασικό ρόλο στο στην διάταξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων που θα αρχίσει να ισχύει ε, το 2016 και ε, καλύπτει τα προσωπικά στοιχεία. Ε, η Κίνα δεν έχει καμία ενισχύ νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Υπό την ισχύουσα νομοθεσία η μεταφορά προσωπικών στοιχείων προς χώρες που δεν εξασφαλίζουν ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας είναι δυνατή μόνο εάν ο εξαγωγέας αυτών των στοιχείων από την Ένωση παρέχει όλες τις ασφάλειες και ασφαλιστικές δικλείδες μέσα στην αστηρή ερμηνεία του κανονισμού. Οι ασφαλιστικές δικλείδες ε, περιλαμβάνουν τη χρήση ε, εργαλείων όπως ε, στάνταρ συμβατικές ρήτρες, ιδιαίτερα όσον αφορά το ναι, σύννεφο, το υπολογιστικό σύννεφο. ενημερώνει και τις, αρχικές, τις εθνικές αρχές εποπτείας δεδομένων που έχουν αρμοδιότητες παρέμβασης. Έχουν την, την αρμοδιότητα να επιβάλλουν το μπλοκάρισμα ενός τμήματος ή το συνόλου των στοιχείων, επίσης να επιβάλλουν ε, περιστασιακή και μόνιμη απαγόρευση της μεταφορές. Η το συνόλο των στοιχειων επισης Ένωση έχει προβεί σε συζητήσεις με την Κίνα στο πλαίσιο του ΑΣΕΑΝ ε, στο, του οποίου είναι μέλος και η Κίνα. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν το διάλογο για να ε, εξηγήσουμε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ε, για να λειτουργήσει αυτή ως επαρκής ασφάλεια για τη μεταφορά ε, των προσωπικών στοιχείων. Όσον αφορά τις απαιτήσει για τον εντοπισμό των στοιχείων, έχουμε τις εθνικές αρχές δημόσιας ασφάλειας που θα πρέπει αυτές να επεκτείνουν την δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων και άρα την ομιμότητα αυτής. Έτσι, εντός, είναι εντός της εντολής της Εποπτικής Αρχής των Κρατών Μελών αρμόδια για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας της οδηγίες περί προστασίας δεδομένων. Η Κίνα έχει οθετήσει διάφορες νομοθεσίε που αφορούν τα κυβερνοασφάλεια και την εθνική ασφάλεια περασμένους 18 μήνες. Η Κομισιόν καλωσόρισε την ευκαιρία να σχολιάσει διάφορες τέτοιε νομοθεσίες και καλωσορίζει την προσπάθεια της Κίνα να βελτιώσει την διαφάνεια στην νομοθετική διαδικασία. Η Κομισιόν έχει καταστήσει σαφές προς την Κίνα ότι η, η, η πολυεθνικές και παγκόσμιες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταφέρουν στοιχεία από τη μία στην άλλη τοποθεσία, αλλά με τις κατάλληλες ασφαλιστικές η, Η κινέζικη ασφάλεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με, ανάλογο, με έναν αναλογικό τρόπο που δεν θα προκαλεί και δεν θα δημιουργεί φραγμού στην αγορά και δεν θα παρεκκλίνει από τις δεσμεύσεις περί ασφάλειας προσωπικών στοιχείων. Ευχαριστώ κύριε Μπούλτς. Ξεκινούν οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Βός έχει το λόγο πρώτα για ένα λεπτό. Κύριε Φως. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όπως αναφέρατε, είμαστε μακριά από ένα πραγματικό επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα των ε, προσώπων σε ό,τι αφορά την Κίνα. Η διαβίβαση λοιπόν προσωπικών δεδομένων προς την Κίνα είναι κάτι παρόλα αυτά το οποίο γίνεται πραγματικότητα μέσω της, του υπολογιστικού νέφους ή μέσω της πλατφόρμας Alibaba στην Κίνα και μια σειρά από ακτιβιστές και άλλοι συνάδελφοι θεωρούν ότι δεν δίδει καμία απόλυτη ασφάλεια αυτή η μορφή διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων όπως έχουμε διαπιστώσει και σε άλλε περιπτώσει με τις ΗΠΑ κτλ. Πώ μπορείτε κυρία Επίτροπε να εξασφαλίσετε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων για τι μεταφορέ δεδομένων που γίνονται ήδη αυτή τη στιγμή προ την Κίνα μπορούν να εξασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων αυτών και πώ μπορούν οι αρμόδιε αρχέ και ο επόπτη για τα προσωπικά δεδομένα που είναι αρμόδιο για τα θέματα αυτά ποιο ρόλο μπορούν να παίξουν για να λειτουργήσει καλύτερα η εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φως. Ο κύριος Μάμικης για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμη κυρία Επίτροπο, αγαπητοί συνάδελφοι. Το νέο μοντέλο προστασία προσωπικών δεδομένων ε, δεν υπάρχει ε, στην Κίνα ακόμη που δεν έχει εφαρμόσει νομοθεσία για τη συλλογή, αποθήκευση, διαβίβαση προσωπικών ε, δεδομένων. Επίσης η Κίνα δεν έχει προσπογράψει καμία συνθήκη με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάτι αντίστοιχο με το πλαίσιο ασφαλούς λιμένα Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ. ΕΕ. Δεν είναι το διεθνώς, διεθνές πρότυπο το ευρωπαϊκό. Ε, είναι άλλα τα όσα ισχύουν στην Ένωση και άλλα στην Κίνα. Στην Κίνα ε, αποδέξει που δεν είναι ένα ιδιώτης, ένας υποκείμενος ε, ε, δεδομένων όπως είναι στην Ένωση, αλλά είναι ένας καταναλωτής. Ναι, δεν υπάρχει καμία κρατική υπηρεσία που θα επιβλέπει ε, την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μόνο έτσι όμως θα μπορούν να προστατευθούν οι ιδιώτες. Ε, τα τελευταία λίγα χρόνια η Κίνα όμως προχώρησε σε κάποια μέτρα, σε κάποια νομικά μέσα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να δοκιμαστεί και να ενισχυθεί αυτή η διαδικασία. Οι εμπορικές σχέσεις σίγουρα ε, θα πρέπει να ενισχυθούν και να μην ε, επηρεαστούν ίσως από την προστασία των δεδομένων, αλλά θα πρέπει η Κίνα να βοηθηθεί και θα πρέπει και η ίδια να δείξει ότι η πρόσφατη προσπάθειά στον τομέα προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα τμήμα ε, της τη της ε, βούλησης να αυτά δεδομένα. Δεν είναι μόνο κάτι μεμονωμένο. Ε, οι συστάσεις ε, έχουν ε, διατυπωθεί με στόχο πρώτον να τηρηθούν οι βασικές αρχές προστασίας δεδομένων, τα δεδομένα, τα δικαιώματα να προστατευθούν για τις διαβάσεις και έχουμε και το μηχανισμό επιβολής. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν να ξεπεράσουν πολλά εμπόδια. Όμως, αν και οι δύο πλευρές γνήσια θέλουν να τα περπηδήσουν τα εμπόδια, θα πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάμικινς. Η κυρία Φαν Στόρκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Συζητούμε σήμερα για τα για την διαβίβαση δεδομένων προς την Κίνα. Εμείς ως Alternative für Deutschland ζητούμε να υπάρξουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους πολίτες και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει και καλύτερη προστασία για την ελεύθερη έκφραση των πολιτών. Η, απόφαση για την περίπτωση Σρέμς του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου της 16 Οκτωβρίου 2015 τονίζει ότι τα δεδομένα, τα προσωπικά και η προστασία τους έχουν μεγάλη σημασία για την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αν οι πολίτες χάσουν την εμπιστοσύνη τους, είδατε τι θέλουν να κάνουν, να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο και έναντι της Κίνας θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ, κύριε Φωνστό. Και ένα λεπτό. Ο κύριος Ζεσκόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι είναι κρίμα που αυτή η ενδιαφέρουσα πολύ επικαιρή συζήτηση μπαίνει τώρα στην μεσιά διάταξη που είναι άδειο το κοινοβούλιο και το ημικύκλιο συγκεκριμένα. Και ούτε και οι δημοσιογράφοι φαίνεται να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Η Τσεχία είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης αναπτύσσει και πολιτικούς και πολιτισμιστικούς ε, δεσμούς. Αυτό συνεπάγεται και περισσότερες διαβιβάσεις δεδομένων, μεταξύ των οποίων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των Ευρωπαϊκών πολιτών. Αυτό κατά την άποψή μου θα μπορούσε δυνητικά να αποβεί επικίνδυνο. Γιατί, επί παραδειγματι, η Κίνα δεν έχει καμία ε, νομοθεσία σε ισχύ, η οποία να άπτεται ε, τη αποθήκευση συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτή η έλλειψη συνιστά κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του πολίτε τη. Επομένω, θα πρέπει, κυρία Επίτροπε, να εξασφαλιστεί ότι οι διαβιβάσει δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα θα ε, διέπονται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό, κύριο Σκέλη η Κομισιόν αναφέρθηκε στον κανονισμό για την προστασία δεδομένων όπως και ο συνάδελφός μου ο κύριος Βος και εγώ υπήρξα εισηγητής για την Επιτροπή Ήτρα για ένα διάστημα τεσσάρων ετών ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθησε βέβαια η κατάσταση με το Safe Harbor που έκλεισε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει αντικατασταθεί από το Privacy Shield. Αλλά έχουμε δείξει μεγάλη χαλαρότητα και αμέλεια σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή δεδομένων με την Κίνα. Συγχρόνως, ξέρουμε ότι αυξάνουν οι ροές δεδομένων προς την Κίνα, χρησιμοποιούνται περισσότερο κινέζικα προϊόντα για το λογισμικό, περισσότερο ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε αυτή την προστασία των δεδομένων, να υπάρξει ένα έδος επέκτασης της ε, Privacy Shield ώστε να καλύψει και τα προϊόντα τα οποία εξάγονται στην Κίνα ή έρχονται από την Κίνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη. Ακολουθεί η διαδικασία ΚΑΣΤΙΑΗ. Ο κύριος Καπούτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Κίνα δεν έχει καμία νομοθεσία που να καλύπτει τη συλλογή, την ε, μεταβίβαση και την ε, κατεργασία προσωπικών στοιχείων και δεν έχει συνάψει καμία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό μοντέλο αποτελεί σημείο αναφορά, αλλά όχι ακόμα παγκοσμίω εφαρμοσμένο ε, προδιαγραφή. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περιορίζει την μεταφορά στοιχείων που δεν σέβονται τις αυστηρές ε, προδιαγραφές σε θέματα ιδιωτικής, ιδιωτικών στοιχείων, ενώ ε, όμως η ανταλλαγή στοιχείων ήδη αποτελεί πραγματικότητα μέσω του cloud computing. Η Κίνα έχει οθετήσει επιθετική εμπορική πολιτική επεκτείνοντας τις ε, ζώνες ελευθέρων συναλλαγών για τους ε, ξένους επενδυτές. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε τι γίνεται με τα στοιχεία των Ευρωπαίων πολιτών και αυτά θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσαμπάσκη επίσης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εμβαθύνει τις εμπορικές της σχέσεις με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Έχουμε έναν κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα που έχει όμως κάποια κενά. Είμαι λίγο επιφυλακτικό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την νομοθεσία μα σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να παρέμουν τα συμφέροντα τρίτων χωρών στη δική μας δουλειά. Δεν θα ήταν συνετό να δώσουμε ελεύθερη πρόσβαση ε, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αν δεν έχουμε εξασφαλίσει επαρκή επίπεδα ασφάλειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσαμπάσκη. Ο κύριο Γιακόφτη για να κλείσει τη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΙ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Οι εμπορικέ μα συναλλαγέ με την Κίνα αυξάνονται και είναι και όλο και πιο πολύπλοκες ε, επιχειρηματικές σχέσεις με μια χώρα που δεν έχει όμως επαρκές σύστημα προστασίας, ε, διατήρησης, ε, αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και εδώ είναι και το πρόβλημα το οποίο δεν θα το αντιμετωπίσουμε ή δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο με την Κίνα αλλά και στις σχέσεις μας με πολλές άλλες χώρες γιατί η προστασία των δεδομένων των πολιτών μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα πρότεινα το εξή. Να μην συζητούμε μόνο ε, τα δεδομένα που πάνε στην Κίνα ε, και ξεχωριστά τα δεδομένα που πάνε στις ΗΠΑ. Και με τους ΗΠΑ και με τους άλλους εταίρους μας καλό θα ήταν πιστεύω να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία έννοια, ένα κόνσεπτ ε, της κυβερνοασφάλειας γενικώ. Αυτό χρειάζεται. Ασφάλιση στον κυβερνοχώρο. Και νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια μαζί με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω και πάλι το λόγο στην κυρία Επίτροπο Μπούλτς. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για τις πολύ χρήσιμες παρεμβάσεις είναι σαφές ότι ο ψηφιακός κόσμος του σήμερα με τις διασυνοριακές ε, ροές είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Τα δικαιώματα των πολιτών πρέπει να προστατευτούν, όπως προβλέπει από το χάρτη και από τη δευτερογενή νομοθεσία. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι απουσία ενδεδειγμένων διαβιβάσεων προσωπικών δεδομένων, οι διαβιβάσει αυτέ θα πρέπει να γίνουν μόνο αν υπάρχουν επαρκή εχέγγυα και ασφαλιστικέ δικλείδε, τι οποίε θα μπορούσαμε να, έχουμε με τι ε, ρήτρε ε, που θα δεσμεύουν ε, του εξαγωγείς και θα αφορούν μεταξύ άλλων μέτρα ασφαλεία, υποχρέωση εφαρμογή τεχνικών οργανωτικών μέτρων για προστασία προσωπικών δεδομένων από δόλια ή ε, εξαμελίας ε, παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημέρωση ε, στα υποκείμενα, στους υποκείμενους δεδομένων, υποχρέωση να επεξεργάζεται τα στοιχεία ο εξαγωγέας κτλ. Και αν υπάρξει εξαμελίας ή δόλια ε, πρόσβαση θα πρέπει να υπάρχει αντιστάθμιση αν υπάρξει ζημία για τον υποκείμενο των δεδομένων. Επίσης, όπως προβλέπει η νομοθεσία, θα πρέπει ο υποκείμενος να μπορεί να επικαλείται τα δικαιώματα τα οποία προβλέπονται σε συμβατικές ρήτρε πριν οι αρχές, ε, ενώπιον των αρχών είτε της χώρας διαμονή του ή της χώρας εγκατάστασης του φορέα του τρίτου κράτου. Σε περίπτωση πολυεθνικών εταιρικών ομίλων θα πρέπει να εφαρμόζονται οι εταιρικοί κανόνες. Αυτό γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται μια ομάδα του ομίλου θα μπορούν ως δικαιούχοι, ε, τρίτη δικαιούχοι να επιβάλλουν την εφαρμογή των κανόνων ενώπιον των αρχών προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να μπορούν να γύρουν αγωγή στα δικαστήρια. Διαβιβάσει δεδομένων με βάση PCR θα πρέπει να εξοδοτούνται από τον DPA, ε, τον, ε, την υπεύθυνη αρχή δηλαδή προστασία δεδομένων για τις χώρες που έχουν ε, μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει το διάλογο με την Κίνα και τους άλλους διεθνείς εταίρους ε, ε, στην Ασία, στη Βόρεια και Νότια Αμερική για την προαγωγή των αρχών που διέπουν την προσέγγιση μας για την προστασία των ροών δεδομένων και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπούλτς. Έχει κλείσει η συζήτηση και για το θέμα της διαβίβασης προσωπικών δεδομένων στην Κίνα. Το